Συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε ήδη φτάσει στις 3 και 10 και είχαμε πει και πρέπει να ξεκινούμε στις 3. Πρώτα απ' όλα θα σας ζητήσω να εγκρίνετε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, δηλαδή αυτή της 14 Νοεμβρίου. να εγκρίνουμε και την ημερήσια διάταξη. Έχετε σχόλια επί της ημερησίας διατάξεως. Όχι από όσο βλέπω. Επομένως προχωρούμε. Η πρώτη έκθεση είναι η έκθεση της κυρίας Λίχτενμπέργκερ για, για τον κανονισμό για στατιστικές σχετικά με τις μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών κτλ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ οι συνάδελφοι οι οποίοι συνέβαλαν δεν είναι ε, στην εργασία μας, ε, δεν ε, έχουν ακόμα φτάσει. Ενώ λέει ομιλήτρια του συναδέλφους που έχουν υποβάλει τροπολογίες, όχι δεν αναφέρομαι στους προέδρους ή τους κοιόδης κτλ. να πω το εξής. Για τις τροπολογίες τις οποίες έχουμε λάβει υπόψη μας, ε, οι περισσότερες με βρίσκουν σύμφωνοι εκτός από ε, αυτές όπου αναφέρεται if needed, εφόσον ε, παραστεί ανάγκη. Ε, αυτό συνήθως μας το λέει το Συμβούλιο, δεν χρειάζεται να το επιβάλλουμε στους εαυτούς μας, επομένως αυτό είναι αρνητικό. Επίσης, τροπολογία Σασάντα για την περίοδο για, για την, κατά την οποία επιτρέπονται η κατεξουσιοδότηση πράξεις Ε, η ε, Κομισιόν σε άλλες περιπτώσεις λέει απεριόριστο χρονικό διάστημα, άλλες λέει 12 μήνες ε, ε, ή 5 χρόνια, συγγνώμη, θα το δούμε, αυτό πρέπει να διορθωθεί. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, ευελπιστώ ότι πρόκειται για ένα θέμα επί του οποίου μπορεί να υπάρξει ευρεία ε, συνένεση. Έχουμε συζητήσει επανειλημμένα για το περιεχόμενο του κανονισμού και της τροποποίησης, επομένως δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε. Ε, δεν ξέρω αν κάποιο ζητά κάποια αποσαφήνιση. Εγώ πάντως από τη δική μου πλευρά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Ε, ούτως ή άλλως μία σκιώδης βρίσκεται εδώ, επομένως θα της δώσω το λόγο αμέσως. Ναι, το όντιμη μόνο εδώ είναι προσαρμογή στη συνθήκη της Λισαβόνας και η συνάδελφος Λίχτεμπερκ ε, βρήκε την ευκαιρία να το προσαρμόσει, να το επαληθεύσει καλύτερα για να δούμε χρειάζεται περισσότερες προσαρμογές. Είναι πολύ σημαντικό. Η ομάδα μου δεν ε, συμφωνεί 100% στον περιορισμό των ε, συμπράξεων. Ε, κατά τα άλλα συμφωνούμε. Απλώς πιστεύω ότι μπορούμε εμείς το Κοινοβούλιο να το βελτιώσουμε. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριο Αρκαντράουι. Έκθεση Λίχτενμπέργκερ, έτσι. Ναι, αυτό ξέρω κύριε Πρόεδρε. Ναι, Πρόεδρε, το ξέρω, το ξέρω. Είμαι ενημέρος. Και ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστώ την Εύα Λίχτενμπέργκερ για τη δουλειά της. Ε, είχα επισημάνει και προηγουμένως που συμφωνούμε για τις προτάσεις αυτές και την προσαρμογή των στατιστικών. Επομένω, είμαστε σύμφωνοι με, τη θέση, με τις θέσεις σου, Εύα. Βεβαίω, μια-δυο τροπολογίε δεν μα βρίσκουν 100% σύμφωνο, αλλά εν γέννη και εν όλο συμφωνούμε. Καλώ είναι ο πρόεδρο, δεν είναι κανεί άλλο εδώ, Εύα. Άρα, επαναλαμβάνουμε ότι αύριο είναι η ψηφοφορία και εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί ο κατάλογος των τροπολογιών ώστε να φαίνεται θετικό πρόσημο από την συγγήτρια για την τροπολογία στις άλλες, τότε θα το πω εγώ πριν από την ψηφοφορία, αλλά φαίνεται ότι έχει ήδη γίνει προσαρμογή. Καλώς, ευχαριστώ και πάμε στο επόμενο θέμα που είναι οι στατιστικές μεταφορών. Τι έχει πει Εύα, θα έρθει, σε έχει ενημερώσει. Ναι, βεβαίως. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ και για τις ε, τροπολογίες σας. Εσύ, εσύ, εσύ, σειρά σου. Ακριβώς, αντί για τον Μίχελ Κράμερ μιλάω εγώ. Γιατί θα αργήσει σήμερα. Ή... να τα πω και γερμανικά καλύτερα. Έχουμε μερικές τροπολογίες και εδώ οι οποίε θέλουν να το where appropriate, όπου αρμόζει. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κατάλληλη λύση, όπως και ο κύριος ε, ε, Κράμερ συμφωνεί άλλωστε, δεν θα πρέπει να περάσει από το Συμβούλιο τους ή άλλους. Και στην ε, τροπολογία Μπόρισοφ, θα ήθελα να επισημάνω ότι θα υπερψηφίσουμε, αλλά, αλλά υπάρχει μια διαφορά ενώ ο κύριο Μπόρισοφ μιλάει για 500 χιλιόμετρα, εμεί έχουμε 500 έως 850 και επιπλέον. Και αυτό είναι λόγω της ανάγκης που βλέπουμε να γίνει διάκριση ε, μεταξύ μεγαλύτερων και μικρότερων κρατών. Να γίνει μια διαφοροποίηση δηλαδή ως προς την ε, ε, έκταση, την επιφάνεια του κράτους. Όλα τα άλλα τα κρίνουμε θετικά. Και συμφωνούμε. Ευχαριστώ Μπόρισοφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Και θα ήθελα να συζητήσουμε τις στατιστικές σχετικές με τα ατυχήματα. Διότι από ό,τι μου φαίνεται θα πρέπει πάντοτε να προσέχουμε να είναι το δικό μας δίκτυο ασφαλές. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται θα πρέπει να είναι δεδομένα ε, σαν τα δεδομένα της Eurostat. Οπότε ίσως δεν θα πρέπει να διαβρύνουμε τόσο πολύ το πεδίο εφαρμογή, ώστε να πάρουμε και δεδομένα από τους δρόμους ε, ή άλλου είδους ε, συνδυασμένες μεταφορές. Θα πρέπει επίσης να μην περιλάβουμε εδώ και στοιχεία σχετικά με τα ποδήλατα. Τώρα όσον αφορά την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τέτοιες κατεξιοδότηση πράξεις είναι γνωστό ότι υπάρχει μια πρόταση ούτω ώστε αυτή η αρμοδιότητα να ισχύει μόνο για πέντε χρόνια ε, τα οποία να επιδέχονται ε, μια παράταση, μια ανανέωση οπότε εγώ είμαι υπέρ των σχετικών προτάσεων όμως θα πρέπει ταυτόχρονα να επιφυλάξουμε για τον εαυτό μας ε, ε της αρμοδιότητας που λέγεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όποτε υπάρχει κατεξοδότηση αρμοδιότητας και επίσης θα πρέπει αντιστέχως <clears throat> να διεξέλθουμε και τα θέματα τα σχετικά με τις συνδρομικές μεταφορές. Συμφωνώ με τον εισηγητή και που λέω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει κάποιες εκθέσεις όπως το λέει ο να έχουμε στατιστικές αν α, ε, ε, μονάδα απόστασης και εγώ όπως και ο συγκητής έχουμε κάποιες ε, αρμοδιότητες συγγνώμη κάποιες τροπολογίες οι οποίες κατέστησαν κατόπιν 20 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριο Σίμψον και τώρα θέλετε να μας πετύχουμε κύριο κύριος Ναι, Πρόεδρε έχω να κάνω μία ε, παρατήρηση ανάλογη με αυτή που έκανα προηγουμένως. Σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με τον εισηγητή, άλλωστε αυτό θα φανεί και από την στάση μας στην αυριανή ψηφοφορία. Αυτό είχα να πω και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Μάισνερ. Ναι, εν γέννη συμφωνώ Νομίζω ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε την πορεία του κειμένου αυτής της έκθεσης. Μία έκθεση λοιπόν, όχι δύο, δεν έχει νόημα να έχουμε δύο. Και χρειάζεται βέβαια και περισσότερη και πιο στενή συνεργασία με τη Eurostat, εξού και τροπολογία υπαριθμών 1. Όπως είπε και το ΕΛΚ, όσο και να μου αρέσει το ποδήλατο, όσο και να συνηθίζω ή να θέλω να μπορώ να φορτώσω το ποδήλατό μου στο τρένο, ίσως είναι υπερβολικό να ασχοληθούμε με την λεπτομέρεια αυτή ε, για την καταγραφή των δεδομένων κατά τη διάρκεια νομίζω της αναθεώρησης του Recast. Η Γενική Διεύθυνση για τις Μεταφορές ε, έκανε μια προσπάθεια με μια βάση δεδομένων ε, που πιστεύω ότι είναι ικανοποιητική. Μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και να ε, βεβαιωθούμε ότι είναι πλήρης και βέβαια με διαφάνεια στην πρόσβαση που είναι και το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Εύα. Κάποιος άλλος. Θες να προσθέσεις μάλλον Εύα κάτι. Έχουμε ένα ρητό στην Αυστρία ότι η στατιστική είναι σκύλος. Σκύλος δηλαδή όχι κάτι το αυθύπαρκτο και με τη δική του αξία, αλλά κάτι το οποίο έχει αξία μόνο εάν προσφέρει υλικό αξιοποιήσιμο. Προσπάθησα, δηλαδή ότι είναι πολύ δύσκολες στατιστικές. Προσπάθησα λοιπόν να δω σε στοιχεία ατυχημάτων για ε, μια φάση ηλικίας από 14 έως 16 και μια άλλη από 16 έως 18. Δεν ήταν συγκρίσιμα τα στοιχεία, δεν ήταν επαρκής η καταγραφή. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ποδήλατα. Άρα από τη μια έχουμε τα ερωτηματικά μας, τη διατύπωση δηλαδή των ζητημάτων που θέλουμε να καλυφθούν από τις στατιστικές, αλλά από την άλλη είναι πράγματα τα οποία ίσως μας ενδιαφέρουν να τα δούμε και σε σχέση με τα πρακτορία μας, τα τουριστικά, για να δούμε τι είδους ε, στατιστικές μπορεί να υπάρχουν για αιτήματα φερρυπίν για ποδήλατα, διότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη προσφορά ε, για ε, επισκέπτες, τουρίστες. Αν ας πούμε σκεφτούμε ότι μπορεί κανείς να κατέβει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Δούναβη στις όχθες του με το ποδήλατο. Έστω μετά μπορεί να δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλά κάποιος που θέλει να κάνει ένα μεγάλο κομμάτι του Δούναβη μέχρι και την Αυστρία ας υποθέσουμε ή και λίγο πιο χαμηλά και μετά να επιστρέψει με το τρένο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει χρησιμότητα ή με το αεροπλάνο. Αυτό έχει σημασία λοιπόν να το δούμε, όπως είπαμε τους πράκτορες, τους τουριστικούς κτλ, που μπορεί να καταγράφεται μια ζήτηση, στη τελευταία ανάλυση είναι αντικείμενο και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και θα ήταν καλό και στην υλοποίηση της νομοθεσίας να είμαστε σε θέση να διευρύνουμε ένα ελκυστικό ε, κάνιστρο προσφορών το οποίο θα αξιοποιηθεί αναλόγως. Και αυτό ίσως ε, μία επιχείρηση να αντίθετα από την τουριστική, το τουριστικό πρακτορείο ή από, τον, από την Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων ε, να μην έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να μην έχει συναντήσει μια τέτοια ζήτηση. Γι' αυτό εμεί ω Κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε θέση να έχουμε μια γενική επισκόπηση του που έχει εμφανιστεί αυτού του τύπου η ζήτηση και που μπορούμε να προσφέρουμε την υπηρεσία. Και επίση, το συγγνώμη για το ότι μακρηγορώ, Μία δυνατότητα για μια προφορική τροπολογία στην υπαριθμόν 19 φαίνεται να έχω σημειώσει, αλλά κατακάλυπτεται και στον κατάλογο των ψηφοφοριών. Συγκεκριμένα στην καταγραφή αριθμό χιλιόμετρων στεροδρομικών υποδομών εξοπλισμένων με το ΕΝΤΕΦ. Θέλω να συμπληρωθεί το μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου που είναι διαρκώς η λέξη διαρκώς δηλαδή, εξοπλισμένο. Γιατί βέβαια αν έχουμε σε κάποια χιλιόμετρα τον εξοπλισμό και σε κάποια άλλα όχι, τότε δεν μας βοηθάει πάρα πολύ. Ε, αλλά όπως είπα θα τον δείτε και στον κατάργο των ψηφοφοριών και σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λίχτενμπέργκερ και που μιλήσατε για ξανά του κύριο Κράμερ. Ε, αύριο θα γίνει η ψηφοφορία. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Είναι του κυρίου Φιλίπ Ντεμπάκερ. Να τον ε, περιμένουμε να έρθει.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 I give you a second to get yourself together because there's no shadows here. Well, I know. Λοιπόν, ε, ε, ε, περιμένουμε σκιώδεις, δεν έχουμε σκιώδεις. Τέλος πάντων, Φίλιπ, είσαι εδώ. Όλοι θα συμφωνήσουν, αφού δεν είναι κανένας εδώ για να πει όχι. Λοιπόν, θα μιλήσω Ολλανδικά καλύτερα. Ε, morgen inderdaad stemmen we over eh, twee dossiers. Λοιπόν, αύριο θα ψηφίσουμε για δύο ε, ζητήματα, ε, δύο φακέλους για αυτό που ονομάζουμε e-call την ανάπτυξη ε, του διαλειτουργικού συστήματος e-call σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ένα δεύτερο ζήτημα που αφορά την ανάπτυξη του συστήματος e-call σε οχήματα. Ε, πιστεύω ότι μαζί με τους σκιώδεις συγητές καταφέραμε να επιτύχουμε καλές συμβιβαστικές λύσεις. Εδώ και καιρό αρχίσαμε να ασχολούμαστε ε, με αυτό το σύστημα του e-call. Είναι κάτι το ε, στο οποίο πιστέψαμε και θελήσαμε να το προχωρήσουμε. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να ε, υπάρξει αυτό το σύστημα e-call. Είναι καλό για όλους τους πολίτες ε, και για τους οδηγούς, γιατί ξέρετε ότι τα πρώτα λεπτά είναι ζωτική σημασίας σε περίπτωση ατυχήματος για τα θύματα με τον τρόπο αυτό ε, θα μπορεί και πιο εύκολα να φτάνουν οι βοήθειες ε, οι οποίες είναι απαραίτητες, θα ανοίγει πιο εύκολα ο δρόμος ή οι υποδομές είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε στο ευρύ κοινό ε, το σύστημα e-call. Ε, βεβαίως ε, θα πρέπει να έχουν και τα κράτη-μέλη την δυνατότητα να φιλτράρουν αυτά τα τηλεφωνήματα που θα γίνονται μέσω του συστήματος e-call έτσι ώστε να μην προκύπτουν εμπλοκές στον αριθμό 112 θα πρέπει να μελετήσουμε ε, το κατά πόσο θα πρέπει αυτό το σύστημα ε, e-call να διευρυνθεί έτσι ώστε να τοποθετηθεί και σε άλλα οχήματα όπως είναι τουριστικά λεωφορεία, σχολικά λεωφορεία, φορτηγά κτλ. Θα πρέπει να ε, υπάρχουν επίσης πλατφόρμες τυποποιημένες επί των οποίων θα μπορούν να εργάζονται ε, ταυτόχρονα ε, πολλοί οργανισμοί πάνω στην ίδια πλατφόρμα. Επίσης ε, ε, κάποιοι έχουν ήδη ε, χρησιμοποιήσει, μάλλον έχουν ήδη αναπτύξει την τεχνολογία του e-call. Οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να υποστούν κυρώσεις. Σημαντικό στοιχείο είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και των εμπιστευτικών στοιχείων. Ε, κατά την άποψή μου, κύριε Πρόεδρε, από την 1η Οκτωβρίου του 2015 θα πρέπει να εξοπλιστούν τα νέα οχήματα με αυτό το e-call γίνεται μια προσπάθεια από ορισμένου να αργοπορήσει αυτή η ε, υποχρέωση. Εγώ αντιθέτω, είμαι τη άποψη ότι θα πρέπει ε, όλοι μαζί να ε, δείξουμε ότι πιστεύουμε ότι πραγματικά θα πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να ισχύσει η υποχρέωση εγκατάστασης του e-call στα νέα οχήματα, να δείξουμε και ένα μήνυμα, να στείλουμε ένα μήνυμα προ το Συμβούλιο ότι είμαστε ενωμένοι. Υπάρχουν βέβαια και πράγματα όπως ε, ε, π.χ. το ενδεχόμενο εξοπλισμού των ε, αγροτικών οχημάτων, τρακτέρ με τον μηχανισμό e Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Κοιτάξτε, πρόκειται για ένα παθητικό σύστημα προστασίας. Δεν θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα γεωεντοπισμού. Επίσης, θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια για την ε, υποχρεωτική τοποθέτηση του e-call ε, στα οχήματα. Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω ότι αύριο το απόγευμα μετά την ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί η συζήτηση για το θέμα αυτό. Κύριε Σκόλ, Κοχ, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σχολούμαι με το θέμα αυτό εδώ και πολλά χρόνια ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την πολύ καλή δουλειά, εισηγητή και σκιώδη εισηγητές. Έχουν νομίζω τα κράτη-μέλη αντιληφθεί ότι πια πρέπει να κάνουν κάτι για να ε, προχωρήσει η κατάσταση και θα πρέπει να διατηρήσουμε τις πιέσεις γιατί χωρίς πίεση βέβαια δεν γίνεται τίποτα. Το έχουμε δει αυτά τα τελευταία χρόνια. Κανείς δεν κινείται χωρίς να του ασκηθούν πίεσεις. Η εισαγωγή στα ε, ιδιωτική χρήση αυτοκίνητα, στα επιβατικά αυτοκίνητα είναι η πρώτη, το πρώτο πιστεύω στάδιο ε, και το απαραίτητο. Δεν χρειάζεται βέβαια απαραίτητα να εισαχθεί σε κάθε τύπου μα με κινητήρα το σύστημα του της ηλεκτρονικής αλλά πάντως οπωσδήποτε σε το χρόνο σε φορτηγά. Ίσως όχι σε τρακτέρ και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ κύριο Σολκαντράου. Ε, ξέρω ότι κύριε Κόμερ έχει, στείλει, έχει πει ότι θα μπορέσει να έρθει. Ευχαριστώ. Εγγνώμη στη Τσίτα της Εσχιώδους Εισηγήτριας να ευχαριστήσω ε, τον εισηγητή για, το, για τη δουλειά του. Ήταν μια μακρά διαδρομή, ούτως ώστε να φτάσουμε στη φάση αυτή ε, της εναρμόνισης για τη διευθυντικη υπηρεσια υπηρεσία e-call και αυτό το 2005 ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα επαναστοξούμε για την ασφάλεια στην Ευρώπη και επομένως ε, έχουμε αυτή την στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια ρυθμιστική διαδικασία ε, και στα δίκτυα επικοινωνίας και στα σημεία απάντησης και τώρα αυτό το περιέλαβε στο πρόγραμμα δράση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μειωθούν οι τραυματισμοί από τα ατυχήματα στην Ευρώπη. Και βεβαίω δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε τώρα όσον αφορά τι τροπολογίε. Βασικά συμφωνούμε με όλε τι τροπολογίε τη κυρία Συνελόβα από την ε, ΙΜΚΟ και από τον εισηγητή, τον κύριο Ντεμπάκερ. Επίση και από του συναδέλφου ε, του ΕΛΚ. Όμω δεν συμφωνούμε τι τροπολογίε που αφορούν ε, αυτού του είδους την ε, ιδιωτική έγκριση για το, για σύστημα γιατί θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε βελτιωμένα πρότυπα. Όσον αφορά αυτό το, το, τα ιδιωτικα συστήματα στήματα e-call τέλος πάντων. Όσον αφορά τα ε, σημεία απάντησης, θέσαμε με κάποιες τροπολογίες και θέλουμε να απορρίψουμε αυτές που θέλουν την αναβολή της προθεσμίας για την εφαρμογή του κανονισμού. Για μας είναι θέμα προτεραιότητας να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα σημεία, τι θα γίνει με τα συστήματα ECOL για το 2015 και όχι για το 2016. Οπότε, εν γέννη θεωρούμε ότι έχει πάρει τη σωστή κατεύθυνση η υπόθεση και ελπίζουμε να είναι ε, βίωνο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αύριο. Κύριε Λίχτενμπεργκερ. Ευχαριστώ. Είναι γνωστό από τις προηγούμενες συστήσεις ότι δεν ε, είμαι ενθουσιώδης υποστήρικτρια του συστήματος αυτού, πάνω απ' όλα γιατί ε, μας το πουλάνε για τους λάθος λόγους. Ε, ατυχήματα δεν μπορεί ούτως ή άλλως να παρεμποδίσει. Μπορεί μόνο να περιορίσει τι συνέπειε ενό ατυχήματο, ε, δηλαδή λίγο πολύ περικοπή του χρόνου διάσωσης. Γι' αυτό εγώ θέλω τουλάχιστον να είμαστε επακριβείς στην ορολογία που χρησιμοποιούμε. Δεν πρόκειται να περιορίσει τα ατυχήματα. Δεν πρόκειται να στείλει να κάνει κάποιο, ε, κάποια παρέμβαση στο σύστημα πέδησης για να φρενάρει το αυτοκίνητο πιο γρήγορα. Το μήνυμα, η γενικά η επικοινωνιακή σας πολιτική είναι πολύ σφαλμένη. Ε, επομένως, η προστασία των δεδομένων είναι πολύ διαφορετικά τα δικά μας μελήματα. Στο 17 έχει πολύ μεγάλη σημασία τροπολογία 17 να γίνει σεβαστή αρχή της ουδετερότητας. Δεν, φανεί, δεν πρέπει να φανεί ότι εμείς υποστηρίζουμε ή ότι ιδρύουμε, εγκαθιδρύουμε μονοπωλιακά συστήματα και μπορώ να σας πω συγκεκριμένα τι εννοώ με ονόματα. Ε, δεν νομίζω ότι εδώ πρέπει να υπάρξει συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκή για την ηλεκτρονική κλίση Βλέπω βέβαια ότι μάλλον θα εισαχθεί με την ε, επιβολή της Βούλης της πλειονοψηφίας. Mm-hmm. Και κάτι ακόμη ότι η διαδικασία της συναπόφασης δεν πρέπει να περισταλεί από την εκτελεστική εξουσίες της Επιτροπής. Ε, δεν θέλω δηλαδή όταν υπάρξει ή αν υπάρξει υπερβολική ε, νομοθετική ρύθμιση για πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να ελέγξουμε νομοθετικά, να ε, έχει φύγει ο έλεγχος από τα χέρια μας ή αν υπάρχουν παράγοντες για τους οποίους χρειάζεται να αξιολογήσουμε αν χρειάζεται η εισαγωγή ενός νέου συστήματος. Φερρυπίν, στον χώρο της γεωργίας ή της δασοκομείας είναι τόσο πιο σοβαρές οι ε, συνέπειες ενός ατυχήματος που ίσως θα είχε νόημα να εξετάσουμε τι δηλήσεις προτείνονται. Από την άλλη πολλά είναι τα μηχανήματα που δεν ε, ε, εξυπηρετούν, δεν καλύπτουν δηλαδή τις ανάγκες. Γι' αυτό αυτό που μας απασχολεί είναι το πόσο εφικτό είναι ένα εισαχθεί σύστημα και ουσιαστικά και στην πρακτική το να έχουμε οι περιοχές, κράτη ολόκληρα με κάποια κεντρικά σημεία επαφής, τηλεφωνικά κέντρα. Θα πρέπει να έχουν αρκετή διάδοση. Μάλιστα νομίζω ότι και η ΙΜΚΟ ή η ΙΝΤΡΑ, μια, μια από τις άλλες επιτροπές μας ε, ε, συζητάει το ίδιο θέμα σχετικά με το νούμερο 12, ο νούμερο της ανάγκης όταν λοιπόν έχουμε γενικά δυσάρεστες αρνητικές εμπειρίες από την ε, κεντρική οργάνωση υπηρεσιών και το γνωρίζω και από τη δική μου την ε, ε, περιφέρεια όπου μπορεί να έρθουν ταυτόχρονα τρία ασθενοφόρα αλλά εάν ακολουθήσει σχετικά σύντομα ένα άλλο ατύχημα δεν είναι κανένα διαθέσιμο για να πάει εκεί. Λοιπόν πρέπει να μας απασχολήσει όλο το ζήτημα του πώς θα γίνει αυτό στην πράξη πώς θα γίνει η κεντρική οργάνωση της, ε, του κέντρου ε, επικοινωνίας, του κέντρου έκτακτης ανάγκης, πώς θα συντονίζει τις εργασίες, γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές έχουν, έχουν εμφανιστεί προβλήματα σε σχέση με το κέντρο επικοινωνίας, έκτακτης ανάγκης και δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα. Και μάλιστα αυτό αφορά πολλές περιοχές, όχι μόνο μία. Επίσης, ε, εάν Φερρυπίν θεωρεί ο οδηγός, ε, ξεκινήσει το σύστημα λειτουργία και θεωρεί ο οδηγός που έχει φτάσει μέχρι τη Ρουμανία ότι υπάρχει και εκεί σύστημα e-call και επαφεθεί σε αυτό. Δεν είναι πολύ πιο επικίνδυνο από το να μην υπάρχει καθόλου. Ε, αυτά πρέπει να τα κοιτάξουμε όλα νομίζω. Προσωπικώς δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να βιαστούμε. Υπάρχουν τεχνολογικές εξελίξεις που μπορούν να μας βοηθήσουν να λύσουμε τα προβλήματα και να προσφέρουμε μέτρα ασφάλειας και σε τεχνολογικό επίπεδο ε, ικανοποιητικά, προηγμένα και ουδέτερα. Με ενδιαφέρει δηλαδή αυτή η τεχνολογική ουδετερότητα. Με ενδιαφέρει να μην το συνεχιματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και... να μην χρειαστεί να ε, περάσει πάρα πολλούς χρόνους για να λύσουμε τα ζητήματα. Ένα εκκρεμέ ζήτημα φερειπίν αυτό των γεωργικών μηχανημάτων θα πρέπει να συζητήσουμε ποια μηχανικά, ε, μηχανήματα γεωργικά θα υπαχθούν και ποια όχι στο σύστημα αυτό. Εν πάση περιπτώσει αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω από τις αρχές που καταγράφονται και για τις συμβαστικές τροπολογίες που ότι συμφωνούμε, αλλά ήθελα να δώσω, ήθελα απλώς να κρούσω ένα, κίνδυνα, ένα κόδωνα κινδύνου για την κατεύθυνση στην οποία πιεζόμαστε. Υπάρχει δουλειά ακόμα να γίνει πριν περάσουμε στη διαδικασία της υλοποίησης. Δεν έχουν λυθεί ακόμη τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ ε, και τον συνάδελφο ε, Μπάκερ για την εργασία και το πνεύμα στο οποίο ε, εργάστηκε. Συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις παρατηρήσεις του. Παρ' όλα αυτά θα κάνω δύο παρατηρήσεις δικές μου μια τροπολογία η οποία θέλει να προτείνει για όσους θέλουν να βάλουν και ένα δεύτερο ε, ε, ε, μπουτόν, ένα δεύτερο κουμπί για την τεχνική βοήθεια έτσι ώστε να υπάρχει ένα, ένας διαχωρισμός των πραγματικών προβλημάτων και αυτών που αφορούν μια τεχνική βλάβη είτε έλλειψη βενζίνης είτε μια λιχνή που έχει καεί ενδεχομένως κτλ. Ε, έχω καταθέσει μια τροπολογία ε, για το πέρασμα από το 2017 στο 2015 Κοιτάξτε, το πρόβλημα, το θέμα δεν είναι να καθυστερήσει η εφαρμογή του μέτρου, γιατί ε, και εγώ συμμερίζομαι τον προβληματισμό των συναδέλφων, ε, αλλά πρέπει να πούμε ότι το ΣΕΠΑΣΕ ε, έχει προβλεφθεί για το 2015. Επομένως, δεν, ε, δεν θα πρέπει να υπάρξει ένα περιθώριο ανάμεσα στην υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος PSAP και ε, της ε, υποχρέωσης των κατασκευαστών να βάζουν στα νέα οχήματα αυτού του είδους το μηχανισμό. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε να αναπτύξουν οι χώρες τα PSAP ε, ε, ε, και μετά να, οι κατασκευαστές να ξεκινήσουν την κατασκευή αυτών των συστημάτων. Γιατί εάν πιέσετε τους πάντες να ξεκινήσουν μαζί φοβούμε ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα. Εάν ξεκινήσουν και οι δύο υποχρεώσεις ταυτόχρονα φοβάμαι ότι θα υπάρξουν επιπλοκές και ενδεχομένως προβληματική εφαρμογή. Επομένως ίσως είναι πιο λογικό πρώτα να λειτουργήσει, να αναπτυχθεί το σύστημα και μετά ε, να ε, αρχίσουμε να επιβάλλουμε στους κατασκευαστές ε, την ενσωμάτωση αυτού του συστήματος στα νέα οχήματα. Επομένως δεν θέλω με κανένα τρόπο να υπάρξει καθυστέρηση ή αργοπορία. Νομίζω απλώς ότι είναι πιο λογικό. Καλό θα ήταν να μην προκύψει οποιαδήποτε σύγχυση. Να υπάρχει η απαραίτητη συνοχή και ο απαραίτητος χρόνος ανάμεσα ε, στην ε, μία εφαρμογή και τη δεύτερη. Ευχαριστώ. Το λόγο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρος. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Να απαντήσω κάποιες από τις ερωτήσεις ε, για να απαντήσω κάποιες παρατηρήσεις και κατόπιν να δώσουμε το λόγο στους αδελφούς από την Γενική για τις επιχειρήσεις. Πρώτα, πρώτα, να απαντήσω στον κύριο Ρικέ. Θα πρέπει να σταθούμε στο ότι ήδη Έχουμε ήδη PSAP και ήδη έχουμε τέτοιου είδου κατανάθεση. Πράξη. Αυτή εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2012. Και σε συνεργασία με τα κρατημέλη έγινε αυτό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που εμείς το κάναμε από μόνοι μας χωρίς να λάβουμε υπόψη κάτι άλλο, χωρίς να λάβουμε υπόψη το, τι θέλουν τα κρατημέλη. Επομένως ε, τελούν εν γνώση αυτής της ε, πράξεως και επίσης έγινε το πρώτο λειτουργική δοκιμή στα πλαίσια του ε, Ευρωπρογράμματος του Euro Project. Επομένως, το θέμα δεν είναι ότι θα έχουμε μια τέτοια νομοθεσία που ε, ξαφνικά αναδύεται από πουθενά. Οπότε, ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει σχέση με τις κλήσεις που δεν είναι κλήσεις ακριβώς ανάγκης. Θέλουμε τα μελη θα πρέπει ελεύθερα να οργανώσουν από μόνα τους ό,τι νομίζουν και να διαπιστώσουν ε, τι μπορούν να οργανώσουν, τι ταιριάζει καλύτερα αναλόγως με ό,τι ισχύει σε αυτά. Επίσης θέλω να πω κάτι άλλο για τη Λίχτεν Λίχτενμπέργκερ όσον αφορά για την, στην κάλυψη. Ξέρουμε ότι αυτό Δηλαδή το e-call πρόκειται να αποδώσει. Και αυτό γιατί το roaming, η περιαγωγή θα πηγαίνει από τον έναν οπερίδρο στον άλλο. Και έτσι θα έχουμε ως ε, βάση το 112. Και κάτι άλλο τώρα στο οποίο θέλω να σταθώ για να επανέλθω είναι ε, τη θέση σε ισχύ της οδηγίας. θεωρούμε ότι ακόμα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, μπορεί να καταφέρουμε και ακόμα επίσης να θεωρούμε ότι θα είναι πάρα πολύ θετικό εάν ε, τηρήσουμε το τεθέν χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Είπατε θα λάβει κάποιος το λόγο από την ε, Γενική Διεύθυνση για τις Επιχειρήσεις. Έχετε το λόγο κύριε μου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όντως από εκεί προέρχομαι από την Γενική των Επιχειρήσεων και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Επιτροπή Μεταφορών και ιδίω τον ε, εισηγητή, τον κύριο Λιμπάκερ για το σχέδιο τη γνωμοδοτήσή του όσον αφορά το σχέδιο κανονισμό και θα ήθελα τώρα να εστιάσω την προσοχή μου σε τρία σημεία τα οποία σήμερα τα συζητήσαμε εδώ και έχουν ε, να κάνουν και με την επιστοπολογία Να ξεκινήσουμε πρώτα πρώτα με το περιφαρμογή τη προτάσεω γιατί όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ξεκάθαρο το περιφαρμογή γιατί προς το παρόν έχουμε κάποιες τροπολογίες που αντιφάσκουν προς αλλήλες. Έχουμε την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αφορά μόνο, μόνο το, το, 112. Το, το e-call 112. Αυτό δηλαδή που έχει να κάνει ε, με τις κλήσεις αυτές της, ε, της ανάγκης. Και υπάρχουν και άλλα σημεία τα οποία θα πρέπει να τα δούμε γιατί δεν έχουν ρυθμιστεί σε αυτόν τον οργανισμό. Επίσης, το το εφαρμογή, αυτό το οποίο ε, συζητήθηκε από διάφορους οι οποίοι το λόγο, ε, να δούμε ποια οχήματα θα καλυφθούν. Προς το παρόν καλύπτονται οι μέτες, τα βαν δηλαδή και τα ε, γιοταχή. Να δούμε όμω τι θα γίνει για να καλύψουμε και τα άλλα οχήματα. Επομένω, αν θέλουμε να παρεκτείνουμε, να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή, τότε δεν θα μπορέσουμε να κινήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα, γιατί θα πρέπει να γίνει και άλλη μελέτη για τα άλλα οχήματα. Και βεβαίω, ε, ακριβώ όπω το προβλέπετε τώρα, όσα λέει αυτή, αυτό το κείμενο, ε, μπορούμε να κάνουμε την επέκταση αυτή στο μέλλον, όπω το έχουμε πει παραπάνω. Αλλά αυτό θα γίνει επί τη βάση λεπτομερούς ενδελεχούς μελέτης και μελέτης των επιπτώσεων και κάποιε μελέτε κόστους κόστους-οφέλους. Κάτι το οποίο ακόμη δεν είναι έτοιμο. Για διάφορους άλλους τύπους οχημάτων τώρα όσον αφορά τον ιδιωτικό βίο και την προστασία των αντιστοίχων δεδομένων Εμεί συμφωνούμε ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει προστασία των δεδομένων και γι' αυτό και στο κείμενο έχουμε αυτές τις συστάσεις του Σώματος Εργασίας του άρθρου 29. Όμως έχουμε κάποιους κανόνες που περιέχονται εδώ στην πρόταση και θα πρέπει με κάποιο άλλο νομοθέτημα να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες. Εμείς έχουμε προτείνει κατά ανάθεση και ε, πράξη και ε, στις τροπολογίες τώρα προτείνεται αυτό να γίνει με τη συνήθινη νομοθετική διαδικασία. Εμείς ε, επισημαίνουμε τους κινδύνους ε, αυτής της πρόβλεψης γιατί αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν να ισχύει το νομοθέτημα χωρίς, τους, ε, χωρίς τη λεπτομερή ρύθμιση. Αυτό το θέλουμε εμείς. Είναι αδύνατον να έχουμε σύνηθες νομοθέτημα ε, έως ότου αρχίσει να ισχύει και στις λεπτομερίες του ρυθμισμένου το πώς θα γίνεται το e-call. Τέλος, όσον αφορά την ε, ημερομηνία θέση ισχύ, συμφωνούμε με τον συνάδελφο γιατί πρόκειται για την οδηγία που έχει το κείμενό μας και πρόκειται για την οδηγία που έχει προτείνει το Κοινοβούλιο στην εκθεσή του Ιδίας Πρωτοβουλίας οπότε είπαμε ότι και εμείς προτείνουμε αυτά τα ίδια προτείνει για το Κοινοβούλιο. Θεωρούμε ότι μέχρι τότε όλα θα είναι έτοιμα για να ε, ισχύσει το νομοθέτημα για, επαναλαμβάνω, για όμως νέα οχήματα και όχι για τα παλαιά. Ο κύριος Ντεμπάκερ. Πρώτα πρώτα, για αυτά τα οποία είπατε, για τα οχήματα. Ο λόγος του μας πρότασή σας είναι διότι όταν βρισκόμαστε σε μια περίπτωση που κάποιος έχει μια ανάγκη και κάποιος έχει μπροστά του δύο κουμπιά, τότε εδώ πέρα υπάρχει ο κίνδυνος της σύγχυσης, γιατί εδώ πέρα υπάρχει να δούμε τι, πώς θα οργανωθεί το PSAP, δηλαδή το κέντρο λήψης με εκπαίδευσης ανάγκης. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα σύστημα που να ισχύει ε, κάποιο φίλτρο και να ξέρουμε τι, τι, τι, κλίση γίνεται. Ε, αυτό νομίζω είναι πιο ενδιαφέρον σαν προσέγγιση. Επίσης είπαμε ε, να μην υπάρχει πίεση προς ε, τα ελαφισμικά όργανα. γιατί αν εμείς έχουμε το περιθώριο καθυστέρηση ε, ενός ή τριών ετών για κάποια τεχνικά ζητήματα, ε, τότε θα πρέπει και τα άλλα θεσμικά όργανα να, να καθυστερήσουν ακόμα παραπάνω. Οπότε αυτό, ε, τι να σου πω, είναι μια προσέγγιση που την, τη μελέτησα. Βεβαίως και ο οδηγός έχει ευθύνη, το είπε και η Δεν είπαμε ότι με αυτό το σύστημα θα σταματήσουν να υπάρχουν τα ατυχήματα. Φυσικά και συνεχίζει να υπάρχει η ευθύνη του οδηγού. Κανεί δεν είπε το αντίθετο. Εάν κάτι συμβεί, απλώ όχι, όχι, κάτι, άλλο είπαμε, τέλος πάντων, παρεξήγησε. Ε, Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, είπαμε ότι εδώ πέρα τις ρήτρε τις έχουμε α, και είπαμε να διατίθενται τα δεδομένα που πρέπει ε, στα PSAP. και με την ανείχνευση να εντοπίζει το πού έγινε το ατύχημα για να μπορεί κάποιο να αντιδράσει, να βοηθήσει. Να υπάρχει συγχρηματοδότηση για αυτά τα ευφυή συστήματα μεταφορών και αυτό. Και πιστεύω ότι τελικά θα υπάρξει ευρία συνένεση γύρω από αυτή την πρόταση. Και μια από το σύστημα αυτό από τεχνολογική πλευρά, τεχνοκρατική πλευρά δουλεύει, να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν. Ο Πρόεδρος αύριο γίνεται η ψηφοφορία. Και σας ευχαριστούμε. Μόνο η κυρία Φώστερ λείπει και θα αρχίσει όλοι οι άλλοι σκέους εδώ. Οπότε πάμε τώρα στο ETS. Ε- ε- ε Ε, οι διεθνεί αεροπορικές μεταφορές του κυρίου Γκρός την έκθεση και μετά γυρίσουμε στην έκθεση του Κάντσιαν στο 7 δηλαδή. Άρα αν, αν δεν διαφωνείτε πάμε στο 8 που είναι η έκθεση σχετική με τις διεθνεί αεροπορικές μεταφορές. Το 8 αντί για το 7. Ευχαριστώ πολύ. Η γνωμοδότηση που έχουμε εδώ ετοιμάσει και υποβάλει έχει προκύψει μέσα από τις συνθήκες που γνωρίζετε. Ε, είχαμε ένα σύστημα stop the clock με το οποίο αποφασίσαμε ότι σε επίπεδο ΙΚΑΟ θα δίναμε τη δυνατότητα τουλάχιστον να αποστέλλονται θετικά μηνύματα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατηρημένη να βρει μια να βοηθήσει στην εξέβρεση μιας παγκόσμιας λύσης και όχι μόνο ευρωπαϊκής. Από την ε, συνεδρίαση λοιπόν αυτή μέχρι τώρα είχα επαφές ε, σε συνάντηση με την Επιτροπή όπου πρέπει με ηλεκτρίνη να πω ότι στη συνάντηση αυτή δεν ήμουν ενήμερος ότι η πρόταση, αυτό το stop the clock δηλαδή, ε, είχε ήδη αρχίσει να προτείνεται να υποκατασταθεί από μια ευρωπαϊκή λύση για τον αέριο χώρο στην Ευρώπη. Και ότι ήταν μάλιστα η εναλλακτική αυτή ήδη στο στάδιο της συζήτησης. Αλλά δεν είχε εξασφαλίσει ε, συμφωνία. Έτσι λοιπόν και σε ε, αντίθεση με τα όσα είχα πει και ε, γραπτά δηλώσει στο παρελθόν, πιστεύω ότι θα ήταν σκόπιμο να έχουμε τη δυνατότητα μέχρι το 2016 να παραταθεί το σύστημα stop the clock, γιατί κανονικά το 2016 ξεκινάει μια, ένας, νέας, ένας νέος γύρος και έχουμε τον όρο ότι η ΙΚΑΟ θα ορίζει προτάσεις ε, για να βρεθεί λύση σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεδομένων λοιπόν όλων αυτών, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί στους διαπραγματευτές ένα περιθώριο διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, stop the clock μέχρι το 2016 και πέραν αυτού, εάν υπάρχει δυνατότητα για μια διμερή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών, δεν θα πρέπει να ε, χάσουμε την ευκαιρία για τη σύναψη μιας τέτοια συμφωνίας. Είναι μια πρόταση που και σε διμερεί διμερείς συναντήσεις με τα κράτη αυτά τα οποία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον έχουμε ήδη προτείνει. Και επίσης και στη συνέχεια εάν το 2016 επεδοϊκάω δεν υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση για τον τρόπο αλλά και το χρονοδιάγραμμα και με χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο τότε να πούμε ότι από το 2016 αυτή η προσέγγιση για τον ενέργειο χώρο Airspace Approach θα περιοριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι χάνουμε πολύ χρόνο στόχο 2016, με την προθεσμία του 2016, αντιθέτω έχουμε περιθώριο για να ρυθμίσουμε κάποιε λεπτομέρειε και να δούμε βεβαίω τι είδου προδιαγραφέ θα βάλουμε για την περίοδο μετά το 2016. Δεν υπάρχει λόγο να πέσουμε στα, στα γόνατα και να παρακαλάμε για ένα διεθνή οργανισμό που θα ρυθμίσει τα θέματα αυτά, εφόσον δεν υπάρχει διάθεση από τα άλλα κράτη, μπορούμε να προχωρήσουμε. Περιμένω να ακούσω τι αντιδράσει των κρατών, των ε, ομάδων, φαντάζομαι ότι θα είναι ανάμεικτε. Πάντως πιστεύω ότι σε μακροπρόθεσμη προοπτική πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε λύσεις και ευρωπαϊκές. Μπορεί κάποιοι να τις θεωρούν προκλητικές, μπορεί κάποιοι να τις θεωρούν λίγες, αλλά πάντως νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η λύση την οποία καταλήγω και περιμένω βεβαίως με πολύ ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις. Ο κύριος Αλκαντράου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την σημαντική εργασία του και τις επεξηγήσεις που μόλις μας έδωσε. Τις τελευταίες 48 ε, ώρες σκέφτηκα πολύ το θέμα αυτό, γιατί έξισα πολύ το κεφάλι μου μέχρι να δω τι θα κάνω, με αυτή, γιατί έλεγε και η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Πρέπει να περιμένουμε μια, από τη μία μεριά λέω, πρέπει να περιμένουμε μια ε, παγκόσμια λύση. Από την άλλη πλευρά η θέση του εισηγητή ε, πηγαίνουν πολύ μακριά. Ε, συμφωνούμε να σταματήσουμε το ρολόι για τώρα και να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διαδικασίες και οι διαπραγματεύσεις. Μέχρι το 2016 θα πρέπει να υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις. Τώρα, μπορούμε να αναρωτηθούμε ε, επί της αρχής αυτού του ε, παγώματος. Αυτό θα πρέπει ε, να σταματήσει το 16 ή να προχωρήσει μέχρι το, να επιμηκυνθεί μέχρι το 2020. Το 2020 για μένα είναι πάρα πολύ μακριά. Δεύτερη παρατήρηση όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής. Δεν ξέρω εάν κατάλαβα καλά ε, και αν ερμήνευσα σωστά τη σκέψη του εισηγητού, αλλά νομίζω ότι ο εισηγητής θέλει να μειώσει το πεδίο εφαρμογής από το 16 και μετά στις ενδοενωσιακές ε, πτήσεις. Δεν αναφέρεται όμως την υπερπτήση ε, του εναερίου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αυτό μπορεί να έχει κυρωτικό αποτέλεσμα. Αναφέρομαι εις τις ε, αρχές διαχείρισης ε, του εναέριου χώρου ε, και τις εταιρείε και τους οργανισμούς οι οποίοι παρακολουθούν τα αεροσκάφη τα οποία εκτελούν υπερπτήσεις αλλά δεν προσγειώνονται. Αυτά τα δύο ζητήματα, η ημερομηνία, το χρονικό περιθώριο δηλαδή και το θέμα των ενδοενεσιακών πτήσεων. Ε, θέλουμε να ξανασκεφτούμε λίγο τα δύο αυτά θέματα τα οποία ανέφερα και θα δούμε τι θα κάνουμε τελικά. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Μπορώ να πω ότι εμείς από την Άλτα υποστηρίζουμε το Ματσιο Γκρόσο. Έχουμε παρατηρήσει δηλαδή ότι αν δεν πάμε να πέσουμε στον τοίχο με το κεφάλι ε, μπορούμε να κερδίσουμε κάπου δεν μπορέσαμε να πείσουμε όλο τον κόσμο, ε, όλα τα κράτη του κόσμου δηλαδή ότι οι δικές μας λύσεις είναι οι καλύτερες. Ε, δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να δώσει λύση σύντομα για μια παγκόσμια λύση κα όπως θα θέλαμε. Αλλά, εν νομίζω ότι οι λύσει ε, του Ματιού Γκρό είναι οι πιο καλέ. Δηλαδή, να συνεχίσουμε με το stop the clock, και να είμαστε έτοιμοι, ε, να έχουμε δηλαδή να κάτσουμε να συζητήσουμε και να αναλογιστούμε τι θα κάνουμε μετά το stop the clock, ουσιαστικά μετά το 2016. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε, τι είδους πίεση μπορούμε να διατηρήσουμε ώστε να βρούμε τελικά, να καταλήξουμε τελικά σε μια παγκόσμια λύση και να αποφύγουμε ταυτόχρονα περιτές ε, περιτά μειονεκτήματα για την ε, αεροπορία των Ευρωπαϊκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, γιατί βέβαια και αυτό είναι απαραίτητο, να μην, βρεθούμε, να μην φέρουμε τη βιομηχανία μας στην αεροπορική σε δυσμενέστερη θέση. Αυτό. Ας ξεκινήσουμε έτσι και να δούμε αναλόγως και πώς θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ κύριε Λίχτενμπέργκερ. Ευχαριστώ όλα αυτά τα θέματα των ε, ανταλλαγών εκπομπών, του συστήματος ανταλλαγών εκπομπών είναι δύσκολα για όλους μας ζητήματα. Καταρχάς δεν είναι εύκολο και να προσαρμοστεί κανείς ε, ή να ε, παρετηθεί από την εφαρμογή του συστήματος μόνο και μόνο γιατί είναι δύσκολο να τηρήσει τις προδιαγραφές. την νικά ό,τι να σας πω δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει ελπίδα για πιο προοδευτική ε, πλειονοψηφία στο εγγύς τουλάχιστον ή ορατό μέλλον. Έχω μιλήσει και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις αμερικανικές των ΗΠΑ, οι οποίες ε, ε, αυτό που μου λένε είναι παρακαλούμε μην προχωράτε με υπερβολικέ απαιτήσει, μην, μην πιέζετε πάρα πολύ να προχωρήσουμε γρήγορα, γιατί και αυτές προσπαθούν από πλευρά τους να αναπτύξουν τις σχετικές πιέσει σε επίπεδο ΗΠΑ και έτσι ξέρουμε ότι μπορούμε εμεί με τη δική μα στάση να επηρεάσουμε τις δυνατότητες, ε, τις ικανότητες δράσεως των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε σχέση σε άλλα κράτη, ε, σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Για, αυτά δηλαδή μπορούν να επιτύχουν στις ε, χώρες τους ώστε να υπάρξει εν τέλει ένα σύστημα στον τομέα αυτόν, ένα σύστημα αποτελεσματικό, ένα σύστημα το οποίο να φέρνει καρπούς και αποτελέσματα. Κατά τα άλλα, και εγώ γνωρίζω πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση, όπως και οι λοιποί συνάδελφοι. Αλλά πρέπει να απευθύνω για άλλη μια φορά έκκληση, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας και απαραίτητο να διατηρήσουμε τις επαφές με τις μη κυβερνητικές αυτές οργανώσεις εκτός Ευρώπης, να επικοινωνούμε μαζί τους και πάντα με ευθύ τρόπο να αναπτύσσουμε και την επικοινωνιακή πολιτική ε, για τα όσα γίνονται εδώ, ώστε και να μην δίνεται η εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναπάβεται και δεν κάνει τίποτα και δεν προχωράει και να προωθούμε την εικόνα της καινοτομίας ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να διατηρήσουμε αυτές τις εποφές, της ε, ανταλλαγές με τους εκπροσώπους των κυβερνητικών οργανώσεων από τρίτα κράτη. Γιατί εάν Φερρυπίν σε ένα-δύο χρόνια εμφανιστεί έστω και μια μηδαμινή ελπίδα για πρόοδο, για κινητικότητα από πλευρά των ΗΠΑ, πρέπει να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και πάνω απ' όλα δεν πρέπει με μια συγκεκριμένη προθεσμία η οποία ενδεχομένως αναβάλλεται επαορίστο, επαορίστο ε, να θέσουμε σε κίνδυνο τις ε, προβλεπόμενες αλλαγές σε μια τρίτη χώρα, ε, προκειμένου τις ΗΠΑ. Άρα πρέπει να διατηρήσουμε τις επαφές με αυτούς τους εταίρους μας, αλλά και να μην καλλιεργήσουμε ένα κλίμα παρέτησης ε, και εγκατάληψης. Η τροπολογία 8 με ενδιαφέρει πολύ. Βλέπω ότι ε, δίνει λύσεις ενδιαφέρουσες, λογικές για διαπραγματεύσεις. Αλλά όπως είπα, έχουμε να αξιολογήσουμε ολόκληρο γαϊτανάκι από προτάσεις οι οποίες μπορούν να, φτάνουν ε, από ε, την πλήρη εγκατάλειψη του συστήματος μέχρι την μεγαλύτερη και εντονότερη ακόμη πίεση πλευράς της Ευρώπης. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι στρατηγικά επί παραδείγματι διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν ε, σε επίπεδο εκπροσώπων ΙΚΑΟ τόσοι πολλοί σύμμαχοι, ούτε καν σε επίπεδο κυβερνήσεων των λοιπόν κρατών, Άρα ίσως θα ήταν σκόπιμο αυτό το μικρό ελάχιστο μηδαμινό μέσον που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην, ε, στον τομέα αυτών να μην το εγκαταλείψουμε τόσο εύκολα. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι ε, υπάρχει κάποιος από την Κομισιόν. Παρατηρήσει εκτός μικροφώνου δεν ακούνε διερμηνείς. Μάτιο. Ναι, ευχαριστώ και σύντομα. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις. Νομίζω ότι συνεννοούμαστε, καταλαβαίνόμαστε και αντιλαμβανόμαστε όλοι τις επιφυλάξεις σημαίνει των ΔΕΝ και ψάχνουμε να βρούμε λύσεις στο δυνατόν πιο αξιόπιστες. Όπως έχει τώρα η πρόταση πάντως πιστεύω και για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, γιατί συμφωνώ ότι θα πρέπει να επιδιώκουμε τις επαφές μαζί τους, μπορεί να αποτελέσει ένα καλό μήνυμα. Βαρσοβία, Φερρυπίνο, που δεν γίνεται τίποτα. Ένα, σε αυτό το δεν έγινε τίποτα στη Βαρσοβία, μπορούμε εμεί να αποστείλουμε ένα σαφέ μήνυμα ότι μπορούμε να είμαστε έτοιμοι το 2016 ή ότι το 2020 μπορούμε να έχουμε και μια σε παγκόσμιο επίπεδο λύση σε λειτουργία. Αυτό νομίζω είναι μια εναλλακτική και νομίζω ότι αποτελεί στοιχείο ισχύω και για τι δύο πλευρέ. και θα πρέπει αναλόγως ε, να κρίνουμε την επιτυχία μας με τα, από τα αποτελέσματα. Αυτό έχω να πω. Εγώ θα προτιμούσα όπως και να είναι το 2015 να είχαμε μια σαφή και συγκεκριμένη λύση, αλλά δεν είναι δεδομένο αυτό. Και έτσι καταθέτω την πρόταση για σαφή ευρωπαϊκή λύση το 2016 ή το 2020 εφόσον μπορεί να έχει έτοιμη μια σε παγκόσμιο επίπεδο λύση η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι εδώ αυτό μπορεί να αποτελέσει και το αντικείμενο της επικοινωνιακής μας πολιτικής και του τρόπου με τον οποίο θα πουλήσουμε το μήνυμά μας προς τα έξω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, 18 Δεκεμβρίου είναι η λίγη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στις 4 το απόγευμα, 16.00. 18 Δεκεμβρίου. Το έγραψε Εύα? Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 16.00, 18 Δεκεμβρίου. Ωραία και η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει την 21η Ιανουαρίου. Πολύ ωραία. Επόμενο θέμα είναι ο ενιαίος ε, ε, ευρωπαϊκός ουρανός. Έφτασε και ο κύριος Μπόλτουιν. Joint Undertaking Opinion to ITRA Πρόκειται για γνωμοδότηση μαζί με την Ήτρε. So, Antonio, you ready to start? Away έχεις το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε προτείνει καμία τροποποίηση. γιατί θεωρούμε ότι ε, στέκει αυτή η ε, αυτό το αίτημα για παράταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Θεωρούμε επίσης ότι πολύ καλά έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα η σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα και επομένως πρέπει να συνεχίσει. Έχουν υποβληθεί πολύ λίγες τροπολογίες. Ε, δεν δέχομαι μονάχα δύο τροπολογίες της συναδέλφου Τικάου. Πρόκειται για τροπολογίες οι οποίες ε, ουσιαστικά αφορούν το γεγονός ότι δεν πρέπει να ε, υπάρξει ε, παράκαμψη της, ε, του δημοσιονομικού κανονισμού και υπάρχει και μια δεύτερη τροπολογία που αφορά την εντολή του εκτελεστικού διευθυντή που θα πρέπει να ισχύσει μέχρι τη 16 Δεκεμβρίου του 2016. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Ευχαριστώ. Everybody's in Christmas mood today, I think. Φαίνεται ότι όλοι περιμένουν τα Χριστούγεννα. Δεν θέλετε να κάνουμε πολλή συζήτηση, θέλετε να τελειώνουμε, εντάξει. Είναι αλήθεια ότι το έχουμε ξανασυζητήσει, η Κομισιόν ε, ε, ζητώ συγγνώμη, δεν είναι ότι δεν φτάσατε στην ώρα σας, εμείς προχωρήσαμε πολύ γρήγορα και ο Σπύρος. Ωραία, κύριε Δανέλη, παρακαλώ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα σε αυτά που ήδη μας είπε ο Αντώνιο οι περισσότερες από τις ε, τροπολογίες που έχει αποδεχτεί ε, υποστηρίζονται για από εμά. Ε, ούτως ή άλλως η, πρόταση της Κομισιόν ήταν εξ αρχής γενικά αποδεχτή από μας. Ευχαριστώ πολύ. κυρία ε, δεν ξέρω βέβαια αν η DG Climate θέλει να παρέμβει πρώτα. Λοιπόν, η κυρία Μάισνερ. Ναι. Προχωράμε όντως πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε προβλέψει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα κάνουμε μια γνωμοδότηση εδώ για το Συμβούλιο. Ορίζον 2020. Πρόκειται για μια πρόταση σημαντική για τους ενιαίους ευρωπαϊκούς ουρανούς, όπως και ο Αντώνιο δεν έχει καταθέσει τροπολογίες έτσι και εγώ. Είναι καλή όμως η πρόταση και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια ενιαία ομοιόμορφη θα έλεγα ψηφοφορία και πλειοψηφία. Τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, για τα άλλα δεν ξέρω, δεσμεύομαι, θα δούμε. Κύριε Μπόλντουιν, βλέπετε τι ε, ε, αρμονία επικρατεί στο Κοινοβούλιο, άρα δεν θα σας ασκηθεί καμία πίεση ο κύριος Μπόλντουιν. Ναι, νομίζω ότι είμαστε όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Θα ζητήσω πάντως από τον συνάδελφο να πάρει το λόγο μάλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να πω ότι και εμείς βεβαίως ε, ε, στηρίζουμε απολύτως ε, την θέση του βουλευτού κυρίου Καντσάν. Πρόκειται για κεντρική σημασίας πρόταση, διότι αφενός διασφαλίζει την επιβίωση και επιμήκυση του Σέζαρα, αλλά ε, γιατί ξεκινάει και έναν νέο κύκλο όσον αφορά ε, το ε, ΣΕΖΑΡ. Πρόκειται για έναν ενάρετο κύκλο, ο οποίος θα πρέπει να συνεχιστεί. Πρόκειται εδώ για έναν πυλώνα, επί του οποίου τα αποτελέσματα είναι συγκεκριμένα, γιατί στα ΦΑΜΣ έχουμε κάποια ζητήματα, ενώ εδώ βλέπουμε απτά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τον κύριο Καντσάν και ευχαριστώ πολύ και όλους. Πάρα πολύ ωραία. Αύριο λοιπόν ε, θα έχουμε την τελική φάση αυτής της ε, αρμονίας που επικρατεί. Λοιπόν, μια και ο εισηγητής είναι ακόμα εδώ, θέλετε μήπως ε, να πείτε δύο λόγια. Θα, θα σας ακούσουμε με πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, μια και ο εισηγητής είναι ακόμα εδώ για το ETS. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ ε, που ε, μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Ίσως είμαι και λίγο λαχανιασμένη γιατί τρέχαμε από το μετρό μέχρι εδώ. Πήγατε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ε, πραγματικά με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε αυτό το ζήτημα γιατί πιστεύουμε ότι είναι προς το συμφέρον όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Ταυτοχρόνως έχουμε την αίσθηση ότι η πρότασή μας και από νομικής και από τεχνικής απόψεως είναι ορθή ε, και ε, μπορούμε να διεκδικήσουμε την ε, συμφωνία. Θεωρούμε ότι οι διατάξεις οι οποίες περιέχονται στην ε, νομοθεσία ε, με, στο μέγιστο δυνατό βαθμό ευθυγραμμίζονται με τις προτάσεις της ΑΙΚΑΟ. Η γνωμοδότηση μιας τρίτης χώρας όμως ε, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να δεσμεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν οι αποφάσεις ε, δεν είναι ε, συγκεκριμένες. Υπάρχει λοιπόν και μια προϋπόθεση κατά αυτή την έννοια έτσι ώστε να υπάρξει ε, συγκεκριμένη πρόοδος ε, εν ώψη του 2020. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ορθή η ενωσιακή πολιτική αλλά και η εφαρμογή της να γίνει με σωστό τρόπο και από άποψη νομοθεσία. Δεν θα πω όμω τίποτα άλλο. Η συζήτηση ούτω ή άλλω από ό,τι καταλαβαίνω ήταν σύντομη αλλά οπωσδήποτε ιδιαίτερα ε, χρήσιμη και φυσικά ειναι αυτό το χρόνο θα συνεχίσει και η ανταλλαγή απόψεων με τους ε, συνομοθέτες. Ε, πάρα πολύ ωραία. Να σας πω λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος, ότι Ολοκληρώσαμε το δημόσιο κομμάτι της συνεδρίασης, θα συνεχίσουμε και κλεισμένο των θυρών γιατί θα έχουμε ενημέρωση σχετικά με τους τριμερείς διαλόγους και μετά θα κάνουμε και ένα διάλειμμα πριν αρχίσει η συνεδρία των συντονιστών. Παρακαλώ πολύ ε, όσοι δεν πρέπει να παρίστανται παρακαλώ πολύ να ε, ε, εγκαταλείψουν την αίθουσα ησύχως γιατί θα συζητήσουμε για τους τριμερείς διαλόγους. If you could clear the room, please, quickly. This does give me an opportunity. Ο πρόεδρος, ε, με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους αρισχέτους κλητήρες, γιατί κάθομαι και θαυμάζω τι